Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι, αντικαθιστώ την κυρία Σόνια Αλφάνο που κολλείεται και δεν θα μπορέσει να έρθει. Ε, έχουμε τη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας μέχρι τις 5.30 και μετά συντονιστές και κλεισμένο το θυρό στην ίδια αίθουσα μετά τις 5.30. Αρχίσουμε ως συνήθως με την έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις να την εγκρίνουμε, λέω, να το εγκρίνουμε. το εγκρίνουμε. Μετά το επόμενο. Επίσκεψη της αντιπροσωπείας Κρίμ στην Σεριβία 16-18 Ιουλίου αποτελούνταν από 10 μέλη και πήγαν στο Βελιγράδι. Συνάντησαν πολλούς παράγοντες και μέλη του Κοινοβουλίου, δικαστικούς, αστυνομικούς, τελωνιακούς, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Τελικά είχαν, πήραν μια εικόνα της χώρας ολόκληρης εν ώψη μάλιστα της ένταξης της στην ένωση και σταθεροποίηση της οικονομίας της μετά από πολλά χρόνια οργανωμένου μπόικοτ εναντίον της. Τα μέλη, ορισμένα από αυτά τα μέλη θα μας περιγράψουν τις εντυπώσεις τους. Μήπως να αρχίσουμε από τον εισηγητή μας τον κύριο Γιακολίνο ή οποιονδήποτε άλλο θέλει να μιλήσει από τα μέλη της αντιπροσωπείας, ο κύριος Νεύτον Ντάν ας πούμε. Αν επιμένετε πρόεδρε. Δεν ζήτησα όντω το λόγο, απλώς ήθελα να πω ότι εγώ ήμουν εκεί τις δύο πρώτες μέρες και μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη και πολύ εντυπωσιακή μας σόκαραν μερικές από αυτά που μας είπαν οι δημοσιογράφοι για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Ένας δημοσιογράφος μας είπε ποια είναι οι συμμορίες που δρούν στη Σερβία είναι η επικεφαλής των ομάδων κρούσης του Μιλόσεβιτς ή επί Μιλόσεβιτς. Και μετά μας είπαν ότι μεγάλο τμήμα του Βελιγραδίου όπου υπάρχουν ωραίες βίλες και μερσεντές και κανείς δεν φαίνεται να δουλεύει είναι γειτονιές όπου ζουν αυτοί οι συμμορείτε και συμμορήτησες. Λυπάμαι λοιπόν πολύ για όλα αυτά και για τη Σερβία γιατί έχουν πολλά προβλήματα πέρα και από τη διαφθορά. Η ε, καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος είναι τεράστιο πυρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σύντομη εντύπωση ο κύριο Ζόντεργκαρντ επίση θέλει να πει κάτι. Και εγώ θα ήθελα σύντομα να σας αναφέρω τις εντυπώσεις μου. Σύμφωνο απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος. Εγώ δύο πράγματα παρατήρησα. Όταν συζητήσαμε με τα τελωνία, συνειδητοποίησαμε ότι ήταν αδύνατο να συλλάβει κανείς το τι συμβαίνει μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου στα σύνορα στην πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα κέντρο διερχομένων για όλων των τύπων της απάτης. Και δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να βάλει τέλος ε, στη διακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων. Και τα τελωνία δεν έχουν φυσικά τα μέσα στη διάθεσή τους για να σταματήσουν όλο αυτό το λαθρεμπόριο. Και άλλοι ίσως να έχουν την ίδια εντύπωση με μένα, δεν ξέρω. Αλλά εμείς επισκεφτήκαμε μια αποθήκη μια αποθήκη όπου όλα τα προϊόντα που είχε κατασχέσει η Σερβική αστυνομία τα πήγαιναν εκεί, αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα. Και όλα αυτά τα αντικείμενα που βρισκόντουσαν σε αυτή την αποθήκη έμπαιναν σε δημοπρασία και το κέρδος των πωλήσεων ήταν υπέρ, ε, ε, υπέρ των πολιτών. Δηλαδή πήγαιναν σε κοινοφελή έργα. Τώρα ε, μερικά από αυτά τα αυτοκίνητα ήταν αυτοκίνητα τεράστιας ε, αξίας. Τα υπόλοιπα ήταν ε, μηχανήματα ψιλικατζίδικα, δηλαδή ηλεκτρονικά παιχνίδια, τέτοια πράγματα, ψιλολογήματα. Ήταν σαν να βρισκόμασταν πραγματικά σε ένα καραβάν σαράι. και είχα την εντύπωση ότι μας έβαλαν για επίδειξη αυτά τα πανάκριβα αυτοκίνητα, μερικά πανάκριβα αυτοκίνητα και μετά όλα τα υπόλοιπα ψηλολογίδια. Αυτό για να μας δείξουν ότι ε, τελικά δεν είναι και τίποτα τρομερή κατάσταση και δεν γίνεται φοβερό εμπόριο. Άλλα σχόλια. Ο κύριος Γιακολίνο, ο εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στη διάρκεια του ταξιδιού καταφέραμε να συλλέξουμε χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να σας θυμίσω ότι πλέον στην Σερβία αναγνωρίζεται πλέον στο έγκλημα σύσταση συμμορίας με μαφιόζικη χρειά. και με τους συναδέλφους καταφέραμε να διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα της εμπορίας ναρκωτικών στην περιοχή και όλα αυτά θα τα βρείτε στο έγγραφό μου. Κυρία Φαγιό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κάτι να προσθέσω μόνο. Λίγα στοιχεία, παρόλο που δεν ε, ήμουν ε, μέλος της αντιπροσωπείας. Πήγα όμως στη Σερβία πριν από τρεις εβδομάδες με την αντιπροσωπεία την άλλη για την νοτιοανατολική Ευρώπη και επιτρέψτε μου να πω μερικά λόγια. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη Σερβία, πέρα από το οργανωμένο έγκλημα και δίπλα από αυτό, που είναι γενικά πρόβλημα της περιοχής, είναι η συστηματική διαφθορά και συστημική διαφθορά. Οι αντιδράσει είναι πολύ καλές γιατί πλέον ο νέος Πρωθυπουργός και ο κύριος Βούτζης είναι ο ε, αρμόδιος υπουργός για αυτά τα θέματα. Έχει ε, θέσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ως στόχο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και διαφθοράς. Και είπαν ότι κανείς δεν θα πρέπει να θεωρεί ότι δεν μπορεί να διωχθεί πλέον. Η κυβέρνηση είναι καινούρια τώρα, δεν έχει συμπληρώσει ούτε 100 μέρες, δεν μπορούμε ακόμα να την κρίνουμε, αλλά ως στόχο έχει την καταπολέμηση της διαφθοράς και από ό,τι ε, φαίνεται έχουν γίνει κάποιες πρόοδοι ε, για την αστυνομική συνεργασία και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αλλά η Σερβία θα πρέπει να κάνει ακόμα περισσότερα Όλοι θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε όλη αυτή την ιστορία είναι το θέμα του κοσυφοπεδίου. Μεγάλη ανεργία, τεράστια εγκληματικότητα, διαφθορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούν οι δύο πλευρές, Σερβίας και Κωσυφοπεδίου, για να υπάρχει ουσιαστική αστυνομική συνεργασία θεσμικής μορφή σε αυτό το επίπεδο για να μπορούν από κοινού να καταποτελούν την ε, εγκληματικότητα και στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Και έρχομαι στη δικαιοσύνη. Και εδώ είναι σημαντική η μεταρρύθμιση της, είναι μακράς πνοή σε αυτός ο στόχος για να υπάρξει ανεξάρτητη δικαιοσύνη στη Σερβία. Χρειάζεται κάποιο χρόνο, αλλά νομίζω ως ε, υποψήφια χώρα προς ένταξη θα επιληφθεί η Σερβία για όλα αυτά τα θέματα. Η κυρία Βάιλερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζω τώρα να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά ε, μου έκανε εντύπωση τα εξή δύο πράγματα ε, στο ταξίδι αυτό. Το πρώτο είναι πόσο ενθουσιώδης είναι οι νέοι, η νέα γενιά και ε, στον τομέα των τελωνίων και στην αστυνομία και με επιτυχίες επισκεφθήκαμε αυτό το πρόγραμμα ε, που ε, δημιουργήθηκε, χτίστηκε ολόκληρο νηπιαγωγείο από το προϊόν εγκλήματος που είχε δημευθεί, κατασχεθεί και ε, αξιοποιηθεί. Βεβαίως η κυβέρνηση μόλις ορκίστηκε και το κοινοβούλιο τώρα έχει εκλεγεί. Χρειάζεται λίγο χρόνο, μερικές εβδομάδες για την υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων. Αυτό φορά ιδιαίτερα ε, το θέμα των δημοσίων ε, προμηθειών, γιατί στο παρελθόν αυτές οι κρατικές προμήθειες ε, ήταν ένα έδαφος για διαφθορά και διαφθορά που έφτανε στο 1 τρίτο, της, το 1 τρίτο του ΑΕΠ. Και τώρα με το νέο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων φιλοδοξούν να είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε ορισμένα σημεία θέλουν να ξεπεράσουν και τις σκανδιναβικές χώρες. Θα δούμε κατά πόσο αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη. Η εφαρμογή καμιά φορά χωλαίνει και φτάνει και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάντως είναι πρόθεση και της κυβέρνησης και της ε, νέας Βουλής όλα αυτά να ισχύσουν και νομίζω ότι είναι ένα πρώτο θετικό μήνυμα. Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσω σύντομες ε, παρατηρήσεις σχετικά με μία εντύπωση που μου διαμορφώθηκε μέσω των επαθών και των πληροφοριών που είχα για τα πιο σημαντικά δηλαδή και πιο ανησυχητικά θέματα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της ε, διαφθοράς. Είναι το πρόβλημα της ανακύκλωσης. Εμείς έχουμε μία χώρα όπου η κουλτούρα της πρόληψης του ελέγχου και της καταπολέμησης της ανακύκλωσης βρίσκεται στα γενοφάσκια του. Εγώ υποστηρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει αυτές τις πλευρές, θα πρέπει να ε, βοηθήσει την, το κυβερνητικό έργο προς αυτήν την κατεύθυνση. Διότι αυτή η χώρα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αύριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να καταστεί ένας παράδεισος ανακυκλωτών με ένα τραπεζικό και ελεγκτικό σύστημα ιδιαίτερα αδύναμα. Πρέπει να τα προσέξουμε αυτά. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο. Άλλες τοποθετήσεις σχετικά. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Τώρα η Σερβία είναι υποψήφια, αλλά Το πρόβλημα είναι να δούμε και με τους συντονιστές τι θα κάνουμε για να συνοδεύσουμε την αντιπροσωπεία. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Επόμενο σημείο. Να τα πω αγγλικά. Διότι εγώ έχω στα αγγλικά το σημείωμά μου. Δεν θα μιλήσουμε για το τέταρτο σημείο. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε γιατί ο εισηγητής μας ο κύριος Γιακολίνο μας ετοίμασε το σχετικό έγγραφο. Ξέρετε ότι η εντολή μας λέει ότι πρέπει να υποβάλουμε μία ενδιάμεση και μία τελική έκθεση. Ο εισηγητής κύριος Γιακολίνο μας είχε πει ότι θα καλύψει τα γενικά, το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος σε τρία χωριστά έγγραφα ένα για το κάθε θέμα και σήμερα θα μας παρουσιάσει το πρώτο τέτοιο έγγραφο με βάση όλα όσα μάθαμε κατά τις ακροάσεις μας και θα μιλήσει σήμερα για το αργανωμένο έγκλημα. Προτείνω λοιπόν η συζήτησή μας να γίνει ως εξής. Πρώτα 20 λεπτά παρουσίαση του εισηγητή, δεν ξέρω αν θα τα χρειαστεί και τα 20 και μετά ένας πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους βουλευτάς. Πρώτα οι συντονιστές και συντονίστριες, μετά τα μέλη. Ο καθένας όμως να περιορίζεται σε δύο λεπτά. Και μετά οι απαντήσεις του εισηγητού. Κύριε Γιακολίνου μου, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. θα κοιτάξω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και συνεκτικός. Μετά από έντονη δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες και με την πολύτιμη βοήθεια πολλών συναδέλφων, συντάξαμε ένα πρώτο έγγραφο εργασίας και με την πολύτιμη βοήθεια της γραμματείας συντάξαμε έλεγα ένα έγγραφο για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την νομιμοποίηση πόρων. Αυτό απαιτεί όμως γνώσεις και ικανότητα για να μπορέσουμε να δείξουμε τις διασυνδέσεις του όλου Προσπαθήσαμε λοιπόν και με, μια, να δώσουμε μια γενική εικόνα με τις διασυνδέσεις του προβλήματος και την κοινωνιολογική προσέγγιση. Και θελήσαμε να δούμε αν η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος είναι ταυτόσιμη σε όλες τις χώρες. Η προβλήματος το έγκλημα σύσταση τιμωρία με, με συνομωτικό χαρακτήρα δεν προβλέπεται από όλα τα κράτη-μέλη. Ορισμένα το έχουν προβλέψει, αλλά αρχίζουν να το συζητάνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να δημιουργήσει μια αστυνομία ικανή να λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για να το κάνει χρειάζεται να έχει τη σχετική νομοθεσία. Το οργανωμένο έγκλημα συνδέεται με διεθνή αδικήματα. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή προσέγγιση και όσο το δυνατόν πιο ευρεία. Δεν υπάρχει ακόμη ορισμός, το λέμε και στην έκθεση. Δεν υπάρχει μια, ένας οικουμενικός ορισμός για το οργανωμένο έγκλημα. Εμείς ψάξαμε να δούμε αν υπάρχουν τέτοιου είδους νομοθετικά μοντέλα σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα. Θεωρήσαμε Θεωρήσαμε ότι είναι οργανωμένο έγκλημα όταν έχουμε μια συμμορία που αποτελείται από πάνω από δύο άτομα και τα οποία εκφοβίζουν για κέρδος, για, να, για, για, για εκφοβισμό και για αποσταθεροποίηση της κοινωνίας. Σήμερα το οργανωμένο έγκλημα είναι πιο ισχυρό από ό,τι στο παρελθόν, έχει εξαπλωθεί γεωγραφικά, έχει καλύψει πολλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και έχει διαρθρωθεί για να διαρκέσει στο χρόνο. Σήμερα εμφανίζεται με επιχειρηματική φυσιογνωμία και διάρθρωση και έχει μολύνει περιοχές οι οποίες στο παρελθόν ούτε μπορείς να το φανταστεί και κανείς και πολιτιστικά και οικονομικά. Το οργανωμένο έγκλημα πουλάει προϊόντα, πουλάει καλά, ε, παράλληλα με την υγιή οικονομία υπάρχει, επιβιώνει και συμβιώνει το οργανωμένο έγκλημα και νόμιμες δραστηριότητες ασκούνται από τις μαθίες. Και παράλληλα έχουμε δραστηριότητες οι οποίες αναγούνται σε αρχές μεθόδους. με τον παραδοσιακό τρόπο διαχείρισης του κέρδους. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις περιοχές εκείνες όπου τα επίπεδα και οι οικονομικές ε, προδιαγραφές είναι ιδιαίτερα υψηλές. Βλέπουμε εμείς να πλήττονται οι περιοχές ναι. που έχουν χαμηλό πολιτιστικό επίπεδο, χαμηλό εκπαιδευτικό σύστημα, νέους, ε, υψηλά ποσοστά ανεργίας και αυτό φυσικά είναι το πεδίο στο οποίο γεννιέται και μεγαλώνει το έγκλημα. Πρέπει λοιπόν εμείς να ενισχύσουμε μια ενιαία προσέγγιση ένα, μια γενικευμένη πρόκληση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Να μπορέσουμε δηλαδή να δραστηριοποιήσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή εισαγγελία. Τα ευρωεγκλήματα χρειάζονται μια συνολική προσέγγιση, μια ευρωπαϊκή εισαγγελία η οποία δεν θα εκτοπίσει τις τοπικές εισαγγελίες αλλά θα συνεργάζεται μαζί τους. Οι μαφίες δρούν σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας. Εμείς έχουμε τέσσερα θεματικά έγγραφα σχετικά με τα διάφορα πεδία σχολιών. Και για αυτά τα τέσσερα έγγραφα θα ήθελα και οι συνάδελφοι που τα συνέταξαν να τα παρουσιάσουν. Ήταν τόσο σημαντική η βοήθειά τους που συμπεριέλαβα τα κείμενά τους στο δικό μου κείμενο. Και η, η Ευρωπόλ μας έχει παρουσιάσει στην ετήσια έκθεσή της ποιοι είναι οι κόμβοι των παρανο... της παράνομης διακίνησης. Και γίνεται και μία αναφορά στον υγιή ε, επιχειρηματικό τομέα, στις υγιείς επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούν αυτές οι μαθίες. Κυρίως αναφέρεται η Νότια Ιταλία ως περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα. Αλλά και τα τελευταία όμως γεγονότα τα οποία έχουμε διαπιστώσει στην Ιταλία, στη Βόρεια και στη Νότια δείχνουν ότι εκεί το, πρόβλημα υφίσταται, αλλά πως υφίσταται και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Είναι Δεν μπορούμε μάλλον σήμερα να πούμε ότι υπάρχει κράτος μέλος το οποίο δεν έχει μαφίες. Αυτό το οποίο έλεγα εισαγωγικά είναι κάτι το υποχρεωτικό πλέον. Περνάμε από λαθρεμπόριο κοσμημάτων σε παράνομες δημοπρασίες, παράνομα στοιχήματα ε, σωματεμπορία, εμπορία, λαθρεμπόριο οργάνων. Έχουμε όλα τα επίπεδα εγκλήματος και όλα αυτά γίνονται με... Ε, ε όλες αυτές οι επιχειρησιακές δραστηριότητες επηρεάζουν την κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στο το περιβάλλον, την εσωτερική αγορά, την υγεία των καταναλωτών βλάπτουν τους ε, τίμιους επιχειρηματίες. και πλήττουν ε, την ε, ειρηνική συμβίωση των κοινωνιών. Μέσα από περίεργες διαπλοκές πολλές φορές εκτόνωσε την οικονομία το οργανωμένο έγκλημα. Πώς μπορεί κανείς όμως να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα εδώ στην Επιτροπή μας με νομοθετικά μέτρα. Μα μερικά είναι φανερά. Εμείς ε, μιλήσαμε για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία την εφαρμογή των ποινών παντού. Κατάσχεση. Το συζητήσανε και στη Λίμπε. Και ο Μίτσελ έκανε και μια έκθεση για την κατάσχεση. Προληπτική κατάσχεση, για παράδειγμα. Κα κατάσχεση πριν από την τελική απόφαση και οι σταστικά δικαστήρια ή για κοινωνικούς λόγους κατάσχεση, δηλαδή αγαθά τα οποία κατάσχουμε από τους μαφιόζους και τα αξιοποιούμε για να καταπολεμήσουμε τη μαφία για δράσεις κοινωνικής ένταξης ή άλλες ε, δραστηριότητες στους ε, δημόσιους, ε, στις δημοπρασίες, στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ας πούμε, ε, δεν μπορούμε να δεχόμαστε εμείς δημοπρασίες από επιχειρήσεις οι οποίες ε, κρατιούνται στα χέρια από τη μαθία για το σώμα τεμπόριο θα πρέπει να μπορέσουμε να θα, θα πρέπει να μπορέσουμε να εκφραστούμε πάνω στο σωματεμπόριο, στο, στη διακίνηση ναρκωτικών. για, το, για το οποία θα μιλήσει ο κύριος ε, Διάς Δεμέρα, είπαμε. Λοιπόν, κατάσχεση, αυστηρή φυλάκιση. Και εμείς σίγουρα θα μιλήσουμε για μερικά πράγματα τα οποία σε συναδέλφους άλλων κρατών μελών μπορούν να, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Εμείς θέλουμε να εμποδίσουμε τους ε, boss, τους gangsters, αυτούς που έχουν καταδικαστεί να σταματήσουν να διαχειρίζονται το έγκλημα μέσα από τη φυλακή. διότι υπάρχει, σίγουρα πρέπει κάποιος να εκτείει την ποινή μέσα σε ένα απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητας. Και σε μια νέα αγορά η εγγύσεις ουσίας θα πρέπει να γίνονται σύμβατα με την ενιαία αγορά και με τον κύριο Ταραμπέλα ε, συζητάμε για το τι μέτρα μπορούμε να φανταστούμε για την, ε, από το να κερδίζουν διαγωνισμούς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταδικαστεί για σύσταση συμμορία στα διάφορα κράτη-μέλη. Μετά, εναρμόνιση και νομοθεσία, της νομοθεσίας των κρατών μελών. Πρόκειται για νομοθετήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουν να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία των εγκληματιών, να ενισχύσουν τους εισαγγελείς, τη χρήση, να ενισχύσουν τη χρήση νέων τεχνολογιών. θα πρέπει να ενισχύσουμε τις νέες ανακριτικές διαδικασίες, να έχουμε μεγαλύτερες ε, τράπεζες ε, δεδομένων. Χωρίς ε, πληροφόρηση δεν μπορούμε εμείς να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης αναφερθήκαμε στην ανάγκη που υπάρχει, και αυτό είναι σημαντικό, να δώσουμε κίνητρα στα κόμματα για την, για την πολιτική τους ευθύνη να δοθεί δηλαδή ένας κατάλογος με αυστηρά κριτήρια, που θα, ένας κώδικας ηθικής που θα εγγυάται την προς ποιος έχει δικαίωμα να αναλαμβάνει σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή, δηλαδή αν έχει, αν είναι, αν έχει εκλογιμότητα, περνώντας δηλαδή και τεστ ηθικού, και ηθικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο των νέων τεχνολογιών, τη χρήση τους. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ένα ψηλό κατόφλι προσοχής. Το οργανωμένο έγκλημα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο, προσαρμόζεται με τρόπο πανεύκολο. Ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, σίγουρα χρειάζεται συμφωνίες με την αστυνομία που είναι συμφωνίες εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών, αλλά χρειάζονται και διμερείς συμφωνίες, ας πούμε Ευρωπαϊκή Ένωση και Βόρειο Αφρικανικές χώρες. Λοιπόν, 17 λεπτά είχα να μιλήσω, τώρα θα ολοκληρώνω μερικά λεπτά, μερικά λεπτά νωρίτερα. Είμαι έτοιμος να ακούσω τους συναδέλφους και περιμένω τις ε, ερωτήσεις για να απαντήσω. Και ευχαριστώ τη Γραμματεία για την πολύτιμη βοήθεια που μου έδωσε. Και πιο συγκεκριμένα τους συναδέλφους που συνέταξαν αυτά τα θεματικά paper, λέει ο μιλητής, τα οποία με βοήθησαν να μιλήσω τόσο ολοκληρωμένα και τόσο διαρθρωμένα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο για την παρουσίασή σας. Μας μιλήσατε για την νομική και την πολιτιστική υπόσταση του φαινομένου της μαφίας και την ανάγκη να δημιουργήσουμε πανευρωπαϊκές πολιτικές. Η κυρία Ματιέ τώρα, εκ μέρους των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ ενθέρμως τον εισηγητή για την Επιτροπή Κρίμα, τον κύριο Γιακολίνο, του οποίου η έκθεση είναι εξαιρετική καθώς και όσους άλλους συμμετέσχουν και θα μιλήσουν και αυτοί για θεματικά τους έγγραφα που προσφέρουν πολλά, προσέφεραν πολλά στη σύνθεση που μας παρουσίασε ο Σαλβατόρε Γιακολίνο. Πράγματι περιγράφει πλήρως το θέμα αρχίζοντας μάλιστα από τον ορισμό του ήταν σημαντικό να υπάρξει και ένας ορισμός σε ενωσιακό επίπεδο του οργανωμένου εγκλήματος και ο ορισμός αυτός είναι πολύ σημαντικός για τη στιγμή που ζούμε σήμερα τουλάχιστον. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα όπως κάνει και εκείνο τη σημασία που έχει η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος ιδίως σε περίοδο κρίσης γιατί οι διάφορες μαφίες μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσονται σε συνθήκες κρίσης με ανησυχητικό ρυθμό και ο εισηγητής μας δίνει ορισμένες διεξόδους για να τις καταπολεμήσουμε. Νομοθετικά μέτρα δηλαδή, γιατί υπάρχει τώρα μια πρόταση της Κομισιόν για την κατάσχεση των εγκληματικών περιουσιών και το αναφέρει και αυτό ο εισηγητής στην εκθεσή του καθώς και το thematic paper του κυρίου Μίτσελ που κάνει και αυτό ορισμένε προτάσεις αλλά επίσης ο εισηγητής αναφέρει τι κάνει η Ιταλία, φέρνει σαν παράδειγμα την Ιταλία για την κατάσχεση των εγκληματικών περιουσιών που θα ήταν και αυτή μία μέθοδος καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Άλλο θεματικό έγγραφο του κυρίου Ντίας Δεμέρα που αναφέρει ακριβώς το θέμα των καρτέλ ναρκωτικών και που δίνει και εκείνο ορισμένες συστάσεις, κάνει ορισμένες συστάσεις και η κυρία Γιάλα Σάντες που μιλάει για το δουλεμπόριο, την εμπορία ανθρώπων δηλαδή και που είναι προφανώς θέμα που αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Η έκθεση λοιπόν αυτή, η πρώτη αυτή έκθεση για το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα μόνο από τρίτο μια πρώτη φάση της όλης ολοκληρωμένης έκθεσης και πρέπει να πω ότι ήδη η πρώτη αυτή φάση είναι πολύ ολοκληρωμένη για την μαφία που είναι ε, σαν ένα καρκίνο στο σώμα της οικονομίας, καρκίνομα και δίνει πολύ ανησυχητικούς αριθμούς και στοιχεία μας δώσατε νομίζω εδώ στοιχεία πολύ πλήρη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εμείς κυρία Ματιού. Είμαι βέβαιος ότι θα προλάβουμε να συζητήσουμε και τα άλλα θεματικά έγγραφα, αλλά αργότερα. Τώρα από τους σοσιαλιστές, ο συντονιστής μήπως. Ευχαριστώ τον κύριο Γιακολίνο για την προσεκτική του δουλειά. Πάω τώρα σημείο προς σημείο. Θέλω να υπογραμμίσω μερικά πράγματα. Πρώτο, η Επιτροπή μας είναι κατά του οργανωμένου εγκλήματος της ε, διαφθοράς νομιμοποίηση πόρων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτός είναι ο τίτλος, γιατί πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες διαπλέκονται μεταξύ τους. Και αυτό το βλέπουμε στην Ιταλία ε, και όχι μόνο στην Ιταλία, ε, μας ε, ανησυχεί ιδιαίτερα για το θέμα της διαφθοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ε, ποιος είναι ο ορισμός του οργανωμένου εγκλήματος. Άμα δεν συμφωνήσουμε με τον ορισμό τότε θα έχουμε προβλήματα και με όλα τα υπόλοιπα. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να μιλήσουμε και για το αδίκημα χορήγησης εκ των έξωθεν βοήθεια. Διότι πρόκειται για εκείνη την γκρι ζώνη, τη θεά ζώνη η οποία είναι η ζώνη, που, η ζώνη των επαφών μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, της πολιτικής, ε, του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμότητας. Τώρα εμείς πολλές φορές ακούμε να μιλάμε εδώ για την Ιταλική μαφία και τις διακλαδώσεις, τις διακλαδώσεις τους στις διάφορες χώρες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό γιατί ναι μεν η Ιταλική μαφία έκανε σχολή. Πρέπει όμως να δούμε και την άλλη την, τοπική εγκληματική ε, ε, οργάνωση η οποία επιτόπου διαμορφώνεται και μετά συνδέεται με την Ιταλική μαφία. Δείτε τι έγινε στη Γερμανία, στο Ντουίσμπουργκ. Δεν είναι μόνο η, η, η, η Ιταλική δράγκετα και οι, οι, οι Καλαβρέζοι οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το έγκλημα. Όχι, πρόκειται για μεταφύτευση μαφιών οι οποίες βρίσκουν έφορο έδαφος και πολλαπλασιάζονται στην επικράτεια. Η κοινωνιολογική πλευρά είναι πολύ σημαντική, αλλά το να το θεωρήσουμε ως υπερισχύον ε, αντικείμενο θα το έβρισκα ε, ιδιαίτερα αφαιρετικό. Εγώ θα θεωρούσα ότι είναι περισσότερο επακόλουθο και όχι προηγούμενο. Η σχέση με την πολιτική είναι από τα πιο σοβαρά θέματα που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και να τα αναπτύξουμε με έναν τρόπο πιο οργανικό και πιο ισχυρό. Μιλήσαμε γι' αυτό στο έγγραφο εργασίας για τη δραστηριότητα με την τοπική αυτοδιοίκηση και έναν ηθικό κώδικα για την διαμόρφωση των ψηφοδελτίων αυτό είναι αφαιρετικό. Δεν είναι μόνο η τοπική αυτοδίκηση η οποία υποφέρει από αυτό. Είναι η πολιτική ιδιαίτερα και η δομή της η οποία δεν εξαρτάται μόνο από το δεν λύνεται, δεν εξαρτάται μόνο η διαφθορά της πολιτικής από πώς είναι διαμορφωμένα τα ψηφοδέλτια πολλές φορές η πολιτική και διαφθείρεται και λειτουργεί υπέρ της ανακύκλωσης. Εσύ μίλησες για την έκθεση της Ευρωπόλ. Πρέπει να τελειώνετε κυρία Μπορτσελίνο. Τελευταία παρατήρηση. Να ρωτήσω γιατί στην έκθεση της Ευρωπόλ μιλάμε για νοτιο ανατολικη ανατολ αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής, Δύσης, Βορρά-Νότου και για την Ιταλία μιλάμε μόνο για, τη, για τον Νότο ενώ θα έπρεπε να πάμε και μέχρι το Μιλάνο που και εκεί έχουμε άλλες πλευρές. Από τους φιλελευθέρους τώρα, ο συνάδελφος Νιούτον Ντάν. Μπίλ, παρακαλώ. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, αξιότιμο εισηγητή του Σαλβατόρου. Έχει κάνει πολλή δουλειά σε ένα τεράστιο ζήτημα. Το πρώτο που είπε είναι το σημαντικότερο. Εμείς σε ποιον αναφερόμαστε, για ποιον γράφουμε αυτές τις εκθέσεις. Γιατί αν ξέρουμε ποιος είναι αποδέκτης θα έχουμε και το ανάλογο περιεχόμενο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αναφερόμαστε ε, στο κοινό που εκπροσωπούμε, που πλήττεται από το έγκλημα και κάνουμε μια σειρά συστάσεων στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν για δράση. Ε, τι μπορεί να διορθωθεί και να πάει καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, για να τον συμφωνήσουμε. Καλή αρχή, λοιπόν, έχει γίνει στο έγγραφο του κυρίου Γιακολίνο. Αυτό που λείπει, βεβαίως, ακόμα λείπουν αρκετά θέματα, είναι η τεράστια μικρή εγκληματικότητα μικρολαθρεμπόριο, παραποιήσεις, προϊόντα μαϊμού, μουσική, ό,τι περνάει τα σύνορα και ε, καταστρέφει πραγματικές θέσεις εργασίας. Αυτό δεν ε, διώκεται ποτέ από την αστυνομία γιατί δεν έχει τους πόρους. Η αστυνομία διώκει τους μεγαλοεγκληματίες, έτσι και τα ηχηρά επεισόδια, γιατί αυτό το πιστώνονται, ε, ο κόσμος φυλακίζεται. Αλλά τι γίνεται με τη μικρή εγκληματικότητα που είναι τεράστια και ποτέ δεν διώκεται, ποτέ δεν υπολογίζεται πουθενά και θα πρέπει να το γράψουμε αυτό. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την αστυνομία να έχει περισσότερους πόρους και χρόνο και χρήματα και διευκολύνσεις για να αντιμετωπίζει κάθε είδος εγκληματικότητας. Γιατί επαναλαμβάνω αυτά τα φαινόμενα καταστρέφουν εκατομμύρια θέσεων εργασία και στερούν από τις κυβερνήσεις μας δισεκατομμύρια. Αυτό ούτε καν το φύγουμε. Χαίρομαι πολύ που βλέπω το τελευταίο παράγραφο 5 το έγγραφο που αρχίζει με τις συστάσεις που μπορούμε να κάνουμε και προσβλέπω στα επόμενα βήματα, στο επόμενο έγγραφο και βεβαίως την κρίσιμη στιγμή για μας είναι όταν θα κάνουμε τροπολογίες όλοι και όλες τις συστάσεις που είμαι βέβαιος ότι όλοι σημειώνουμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο τελικό έγγραφο που φοβάμαι θα είναι και αρκετά ογκώδες. Πάντως, Σαλβατόρε, μπράβο σου, καλή αρχή έκανες και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω Εάν από τους πρασίνους θέλει κανείς να μιλήσει, δεν ζητεί το λόγο κανείς, όχι. Νικόλ, η κυρία Κερνιένσεν, παρακαλώ. Merci. Je voulais juste euh, dire un mot. Ευχαριστώ μια λέξη μόνο. Ή δύο λόγια. Για μια πτυχή της εγκληματικότητας που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είμαι μέλος της Επιτροπής Γυναικών και Πράγματι το δουλεμπόριο ή το εμπόριο ανθρώπων, ιδιαίτερα δε γυναικών, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αναρωτιέμαι αν δεν πρέπει να συνδέσουμε το θέμα της νομοθεσίας για την πορνεία που υπάρχει για πολλές φορές μέλη με τα δικά μας θέματα. Είναι και αυτό μια πτυχή που θα ήθελα να συζητηθεί. Ευχαριστούμε. Από τους συντηρητικούς, για τους συντηρητικούς, κυρία Κλά. Ευχαριστώ. Επειδή διάβασα τα έγγραφα αυτά, καταλαβαίνω ότι το συμπέρασμά μου μάλλον είναι ότι χρειάζεται να συνδυάσουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα και μέσα σε ολόκληρη την Ένωση και διεθνώς και να βρούμε ένα μηχανισμό τις πληροφορίες αυτές να τις διαδώσουμε. Και αφού διαδοθούν να γίνει και κάτι για όλα αυτά, για να φαίνεται, να φανεί ότι κάνουμε κάτι για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να υποστηρίξουμε τις οργανώσεις και υπηρεσίες που καταπολεμούν το οργανωμένο έγκλημα. γιατί οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών αυτών καταπολέμησης κοστίζουν πολύ και πρέπει να τις βοηθήσουμε πρώτον και δεύτερον να κάνουμε μια επιμόρφωση του κόσμου, πληροφόρηση, τι είναι ή το οργανωμένο έγκλημα τύπου μαφίας και ποιες είναι και οι νέες μορφές του όπως το κυβερνοέγκλημα. Ευχαριστούμε κυρία Μακλάρκιν. Τώρα εξ ονόματος της Γκουε για την Γκουε ο κύριος Σόνεγκος. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για το έργο του που είναι τεράστιο και πολύ σημαντικό και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα ήθελα όμως να μιλήσω για ορισμένες ελλείψεις που βλέπω. Ιδίω αν θέλουμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στη σελίδα 4 ο εισηγητής και τονίζει και δίκαια ποια είναι, ποιες είναι οι κοινωνικές πτυχές που καταλήγουν στο έγκλημα όπως η ανέχεια και τα λοιπά. Αλλά στο συμπέρασμά του δεν λέει τίποτα ως προς αυτές τις παρατηρήσεις που είναι πολύ συγκεκριμένες και σωστές μου φαίνεται. Αν έχουμε ως στόχο να κάνουμε προτάσεις κατά πολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να λείπει αυτό το στοιχείο. Να βγάλετε και συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις σας αυτές δηλαδή. Να μας πείτε τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα. Άλλο παράδειγμα ανάλογο. Ο εισηγητής στη σελίδα 6 μιλάει και δικαίως, παρατηρεί μάλλον, ότι η σημερινή κρίση έχει αυξήσει τις δυνατότητες εγκληματικών δραστηριοτήτων, οικονομικών εγκληματικών δραστηριοτήτων και μας λέει ότι λόγω του προβλήματος της δυσκολίας χορήγησης ή δανείων από τις τράπεζες υπάρχει κάτι που διευκολύνει εδώ το οργανωμένο έγκλημα αλλά το συμπέρασμα ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτό. Πολύ σωστές είναι οι παρατηρήσεις σας, αλλά δεν βγάζετε συμπέρασμα. Άλλο σημείο που μου φαίνεται σημαντικό και που δεν βρίσκεται στις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να δώσετε μεγαλύτερη σημασία στο ρόλο της απορρίθμισης του τραπεζικού τομέα, της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων Σήμερα υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για εγκληματική δραστηριότητα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια κεφάλαια που διακινεί το οργανωμένο έγκλημα και στην Ανατολική Ευρώπη και εδώ και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά διευκολύνονται από την απορρίθμιση και είναι αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο που δεν εμφανίζεται πουθενά ούτε ως παρατήρηση ούτε ως συμπέρασμα. Εδώ λοιπόν για μένα τι λείπει στην έκθεση αυτή που περιέχει εξαιρετικές παρατηρήσεις και ευχαριστώ ακόμη μια φορά τον εισηγητή, ελπίζω δεν να συμπεριλάβει και αυτά στις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε και για ο κύριος Μολγκασί τώρα για την ομάδα του. Εγώ συμφωνώ, λέει ο κύριος Μποργκέτσιο με όλους τους επένους για αυτήν την τόσο ολοκληρωμένη έκθεση. Δύο σημεία εγώ θέλω να υπογραμμίξω. Παρακολούθηση και συνείδηση της επικινδυνότητας των μαφιόζικων κεφαλαίων που μολύνουν την κανονική οικονομία και σε μία φάση κρίσης και σκεφτείτε δηλαδή και με την πλαστογραφία τι γίνεται δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο και μια άλλη στάση πολιτικού θάρρους είναι η υπογράμμιση του ρόλου του οργανωμένου εγκλήματος στο σωματεμπόριο και στη λαθρομετανάστευση. Πρόκειται για ένα ταμπού που πολιτικό ταμπού το οποίο ε, πήραζε πολλές ευαισθησίες Όλοι οι πνιγμοί στα σαπιοκάραβα που διασχίζουν την Μεσόγειο είναι πνιγμοί που οφείλονται στο οργανωμένο έγκλημα και στη δράση του. Πρέπει όλοι να λάβουν υπόψη την ανάγκη ότι πρέπει να εγκριζώσουμε αυτά τα φαινόμενα. Τελευταία παρατήρηση γενικού χαρακτήρα. Πολύ καλά έκανε ο εξαιρετικός μας εισηγητής να δώσει ένα πλαίσιο μέτρων για την καταπολέμηση εξπόστε εκ των υστέρων. Αλλά με τη δική μας την Ιταλική εμπειρία, το βλέπουμε δηλαδή αυτούς τους τελευταίους μήνες, περιοχές όπως η Βόρεια Ιταλία, που παραδοσιακά δεν είχαμε τη μαφία εκεί πάνω. Σήμερα βλέπουμε ε, εντυπωσιακή παρουσία των ε, του οργανωμένου εγκλήματος και το ίδιο ισχύει και για όλη την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να πάρει κανείς παράδειγμα μόνο το πώς υπήρξε δίσδυση της μαφίας στις περιοχές εκείνες που προσπάθησε η Ιταλία να τις κρατήσει αμόλυντες με πρόληψη πρόληψη της δίσδυσης αυτού του ιού πρόκειται για πραγματικό ιό ο οποίος λειτουργεί εγκληματικά, οικονομικά αλλά και πολιτιστικά. Γιατί φαντάζομαι ότι για ορισμένες χώρες που δεν είναι όμορες με την Ιταλία, η γνώση που έχουν για τη μαφία και η εμπειρία είναι τα φιλμ του Κόπολα. Και υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση για την πραγματικότητα, για την επικινδυνότητα και για τη δυνατότητα της μαφίας να δυσδύει σε όλους τους τομείς, και στον πολιτικό και στον πολιτιστικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε αυτό το οποίο συνέβη σε ορισμένες βόρειες περιοχές της χώρας μας να γίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τελειώσαμε με τις πολιτικές ομάδες. Κέλλερ και μετά η άλλα Σέντερ. Δύο λεπτά ο καθένας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή δεν θέλω να σχολιάσω, λέει ο κύριο Έλερ, να συμπληρώσω. Είμαι ένα από τους δύο εισηγητέ για το πρόγραμμα έρευνας για την ασφάλεια και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα. Το Κοινοβούλιο στο πρόγραμμα ε, πλαίσιο για την έρευνα ζήτησε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ να εγγραφούν για την έρευνα ασφαλείας για συγκεκριμένε αποστολέ, όχι γενική έρευνα και μέχρι και τις προμήθειε φτάνει αυτό το κονδύλι. Είναι σημαντικό για την Ευρωπόλ να γνωρίζουμε ότι σήμερα από τα κονδύλια αυτά δεν δίνονται χρήματα στη Ευρωπόλ. Δηλαδή το Κοινοβούλιο ζητάει για το κέντρο του κυβερνοχώρου να δώσουμε συγκεκριμένα κονδύλια σε γραμμή προπολογισμού. Και θα ήθελα να πω το εξή, το πιο απευθυνόμαστε ε, δεν θα το απαντήσουν κάποιοι τρίτοι, αλλά μπορούμε να το απαντήσουμε εμεί. Τι κάνουμε εμεί, πώς διαχειριζόμαστε τα κονδύλια και πώς τα εγγράφουμε στον προπολογισμό. Δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα, και η Europol και η Eurojust μπορεί από το κονδύλι αυτό στον ορίζοντα 2020 να χρηματοδοτούνται. Έχουμε μια αποστολή για την ασφάλεια στο χώρο της τάξης των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα όμως, από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα στο κέντρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το ίδιο ισχύει για τράπεζες δεδομένων, το ίδιο ισχύει ε, για βάσεις δεδομένων και για ε, δημιουργία τεχνικών δομών ε, για την καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εδώ να φτιάξω μια γέφυρα ε, με τις ίδιες ε, αποστολές και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Κοινοβουλίου, ότι πολλά από αυτά τα θέματα μπορούμε να τα συνοδεύουμε και με παρατηρήσεις για οικονομικούς πόρους ε, δηλαδή να μην απευθυνόμαστε μόνο σε τρίτους, στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να λέμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ τώρα η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαι εισηγήτρια για το θεματικό έγγραφο για ε, το δουλεμπόριο ε, και το τράφικινγκ και υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα, ας πούμε η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών που δυστυχώς αυξάνεται, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εκμετάλλευση στους εργασιακούς χώρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή για την έκθεσή του και για τον κόπο του και για την προθυμία του να μας ακούει αυτούς που εργαζόμαστε παράλληλα για να ε, βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας ε, στα συμπεράσματα του εγγράφου και ακριβώς πιο που μιλάω στα συμπεράσματα, τα πρώτα συμπεράσματα να πω τα εξή δύο, να σχολιάσω. Ε, στο οικονομικό σκέλος όταν ε, κάνει λόγο για ε, την κατάσχεση και μόνο. Μα αυτό είναι το τέλος του δρόμου και της διαδικασίας. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ενισχύσουμε με πάρα πολύ σαφή και ξεκάθαρο τρόπο την ανείχνευση των χρημάτων πριν φτάσουμε στην κατάσχεση. Δηλαδή, τι εννοώ, σε ό,τι αφορά το τράφικινγκ, αυτό το, τη διακίνηση ανθρώπων ακούμε τις μαρτυρίες, οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται πιέσει και είναι σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση, αλλά τα χρήματα, ε, όπως είπε κύριος Έλε, θα πρέπει να εντοπίζονται εκ των προτέρων. Δηλαδή, πώς διακινούνται αυτά τα λεφτά, εν πάση ακόμα και πριν τη μετακίνησή τους, ε, με κάποιες επιχειρήσεις, εταιρείες που χρηματοδοτούν άλλε δραστηριότητε. Αυτό που μα ενδιαφέρει λοιπόν δεν είναι μόνο η κατάσχεση του προϊόντο εγκλήματο, αλλά να ενισχύσουμε την ανείχνευση ε, των διαδρομών του για να μπορέσουμε να φτάσουμε και σε άλλα χωράφια, γιατί απαιτούμε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και αλλού, και στις φορολογικούς παραδείσους και κάποια άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το ξέπλυμα. Ε, και τώρα, η οριστική καταδίκη. Ο κύριος ε, Γιακολίνο λογικά ε, κάνει λόγο για την τελεσίδικη καταδίκη. γιατί την ε, να μην μπορεί να εκλέγεται κάποιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή να μην συμμετέχει ε, σε διαγωνισμούς. Ναι, αλλά πόσο θα είναι αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι πόσα χρόνια, γιατί πολλές φορές το οργανωμένο έγκλημα το υπολογίζουν και αυτό, ότι θα πάρει τόσο χρόνο η διαδικασία και η δίκη ώστε του συμφέρει. Δηλαδή, να μην πούμε για οριστική καταδίκη, αλλά ακόμα από το γεγονός της υποψίας, αν υπάρχουν αποχρόντες λόγοι ε, να υπάρχουν κάποιες βάσιμες υποψίες, να μην συμμετέχουν ε, ούτε σε διαγωνισμούς, ούτε να μπορούν να εκλέγονται. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής τώρα για να ολοκληρώσει ο κύριος Γιακολίνο. Παρακαλώ μην υπερβείτε το τετράλεπτο και να απαντήσετε στα σχόλια του συναδέλφων. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω, Πρόεδρε. πολλές ε, και ωραίες τοποθετήσεις. Εδώ έχω ένα πρώτο έγγραφο εργασίας. Και η Αγιάλα Σέντερ αλλά και άλλοι αναφέρθηκαν σε ζητήματα οικονομικού χαρακτήρα. Εμείς όμως σήμερα μιλάμε για ένα προσχέδιο για ένα πρώτο έγγραφο. Μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και έκθεση για την ανακύκλωση. Και σίγουρα θα είναι πιο αναλυτικά εκεί ε, όλα τα στοιχεία. Το θέμα της ανείχνευσης, το θέμα της κατάσχεσης, το θέμα λοιπόν της ανακύκλωσης, όλα αυτά θα εξεταστούν. Συμφωνώ ότι και Ευρωπόλ και Eurojust πρέπει να έχουν περισσότερα κονδύλια. Και εγώ το είπα και... Το είπα για τον προϋπολογισμό. Τώρα η κρίση πρόσβασης στη δανειοδότηση είναι κάτι το οποίο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωράει στην ε, Τραπεζική Ένωση γιατί και σε διεθνές επίπεδο να μην γίνει κάτι τέτοιο. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Μποργέτσιο για την επικινδυνότητα των μαφιών ε, και για αυτά που είπε η κυρία Μπορσελίνο έχει δίκιο. Αλλά το θέμα της παροχής εκ των έξωθεν βοήθεια ε, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ας λύσουμε πρώτα το θέμα της σύστασης συμμορίας σε νομοθετικό επίπεδο ε, στην Ευρώπη. Η συνάδελφος Ματιέ πολύ ωραία μας τα είπε. Και έχουμε μία εξαιρετική ευκαιρία. Το θέμα της ε, μη εκλογιμότητας δεν πρέπει να συνδέεται μόνο με την ρες judicata, με τη διδικασμένη πράξη. πρέπει πρέπει ακόμη και αν τα αδικήματα δεν έχουν τιμωρηθεί εν αναμονή αυτής της απόφασης, ο υποψήφιος δεν θα πρέπει δικαίωμα να, να έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα ισχυρό που θα στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι όλα όσα υπόθηκαν θα αποκτήσουν νόημα όταν έχουμε μία συγκροτημένη πλέον δομή της έκθεσης και προχωρήσουμε στις τροπολογίες. Και όπως έλεγε ο Νιούτον Ντάν, να κατεστεί αυτό το κείμενο ένα σημείο αναφοράς για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ τον Σαλβατόρε Γιατκολίνο, τον εισηγητή και όλους όσους συμμετείχαν στο πρώτο τμήμα της συζήτησης. Πάμε στο επόμενο σημείο με δύο θεματικά Ε, και θα περάσω στα αγγλικά. Όπως γνωρίζετε έχουμε τέσσερα θεματικά έγγραφα τώρα για το οργανωμένο έγκλημα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση από το θέμα αυτό. Ε, τα θεματικά έγγραφα έχετε τα γνωρίζετε, τα έχετε ήδη δει Μερικά από τα στοιχεία αυτά τα έχει ήδη συμπεριλάβει στην έκθεση του κύριο Γιακολίνο, αλλά θα εμβαθύνουμε τώρα στη ζήτηση με τους ε, συγητέ μας. Έχουμε για τα καρτέλ ναρκωτικών και τη ε, διασύνδεσή τους με το ε, Ευρωπαϊκό Οργανωμένο Έγκλημα του κυρίου Ντία Δεμέρα, κατάσχεση και δίνημευση προϊόντων εγκλήματος, είναι του Γκέι Μίτσελ Έχουμε στη συνέχεια ένα θεματικό έγγραφο για το τράφικινγκ, διακίνηση ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της κυρίας Αγιάλα. Και επίση ένα άλλο τελευταίο, χωρί να είναι το λιγότερο σημαντικό βέβαια, ε, το κυβερνοέγκλημα. Νέες στρατηγικές έρευνα και νέες τεχνολογίες τη συναδέλφου Έμα Μακλάρκιν. Δεν είναι παρόντε στην αίθουσα ε, όλοι οι συνάδελφοι που έχουν εκπονήσει τα έγγραφα. Θα αρχίσουμε από τους παρόντες, έκαστος ένα πεντάλεπτο για να παρουσιάσει το κείμενό του και υποθέτω θα έρθουν και οι υπόλοιποι όσοι απουσιάζουν στο μεταξύ για να μας παρουσιάσουν την έκθεσή του ο καθένας και θα ακολουθήσει η συζήτηση ε, δύο λεπτά η κάθε τοποθέτηση και θα απαντήσουν οι συντάκτες επειδή θα συζητήσουμε ταυτόχρονα και τα τέσσερα έγγραφα, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους αν έχετε να κάνετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, σε ποιον απευθύνεστε να μας λέτε κάθε φορά. Γιατί θα ζητήσουμε και τα τέσσερα έγγραφα ταυτόχρονα. Ωραία. Προτείνω να αρχίσουμε από τον κύριο Ντίας Δεμέρα. Τα καρτέλ των ναρκωτικών και οι σχέσεις τους με το ε, Ευρωπαϊκό Οργανωμένο Έγκλημα. Έχει το λόγο, αγαπητέ Αγουστή Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε, όπως ε, είπατε και εσείς, το θεματικό μου έγγραφο για τα καρτέλ των ναρκωτικών και τις διασυνδέσεις που έχουμε το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουν τι είναι καρτέλ το καρτέλ είναι μια εγκληματική οργάνωση που έχει ως στόχο την προώθηση και τον ε, έλεγχο ε, διακίνησης ναρκωτικών. Με ποιο στόχο? Με στόχο να επηρεάσει την παραγωγή και τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών. Αυτά τα καρτέλ βρίσκονται κυρίως στην Κολομβία, Γουατεμάλα, Ονδούρα και Σαλβαδόρ Τρινιντάτ και τον Πάγο, στη Δομινικανή ε, Δημοκρατία, στο Μεξικό, στο Μεξικό, συγγνώμη, Αφγανιστάν, Πακιστάν και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Πολλά από τα καρτέλα αυτά συνεργάζονται μεταξύ τους δε. Στη Λατινική Αμερική Γνωρίζουμε ότι είναι ε, πολύ γνωστές αυτές οι οργανώσεις του κοινού εγκλήματος, συνεργάζονται και με ευρωπαϊκές οργανώσεις και στη Λατινική Αμερική έχουν σχέση και με την κυριότητα και με την απάτη, πλαστογραφία, διακίνηση ανθρώπων, παραχάραξη, ξέπλυμα χρήματο, λαθεμπόριο όπλων, απαγωγές και παράνομη κράτηση ε, διαφόρων προσώπων. Θα πρέπει όμως να σας πω ότι το σημαντικότερο ε, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων ε, ως εμπορική δραστηριότητα και εγκληματική είναι η διακίνηση κοκαίνης την Κολομβία, το Περού και τη Βολιβία είναι αυτές ε, οι ομάδες και παραστρατιωτικές μάλιστα και τρομοκρατικές που ελέγχουν την παραγωγή και την ε, διακίνηση κοκαΐνης. Ε, ταυτόχρονα συνεργάζονται με αντάρτες και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις τη μία κατηγορία χωρίς την άλλη. Οι εγκληματίες στην Κολομβία ελέγχουν την κοκαΐνη και συνεργάζονται με άλλες μορφές εγκλήματος στην Ευρώπη. Όπως γνωρίζετε για την κοκαίνη είναι ο δεύτερος ε, παγκόσμιος καταναλωτής κοκαίνης η Ευρώπη μετά τις Ηνωμένε Πολιτείες. Η διακίνηση κοκαίνης αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Όλα, ανεξαιρέτως. Και αυτό βεβαίως είναι συνέπεια μιας διεθνούς οργάνωσης με ε, αλυσίδα από την παραγωγή στην κατανάλωση θα λέγαμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η μητέρα όλων αυτών των ιστοριών είναι ε, ομάδες από τη Λατινική Αμερική. Τι συμβαίνει όμως. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες ε, και συντονισμένες Ευρώπης, Λατινικής Αμερικής για την καταστολή αυτών των ομάδων. Οπότε αυτές οι ομάδες μετακινούνται. Όπου καταστέλλονται σηκώνονται και φεύγουν. Δεν έχουν καμία έδρα γεωγραφική, ε, ούτε πρόβλημα χρόνου να μετακινούνται τα σύνορα Βενεζουέλας η ε, σημερινού ε, βλέπουν μαζική ε, εξαγωγή αυτού του προϊόντος και διαθαλάσσεις και αέρος γίνεται η μεταφορά. Τώρα για το Μεξικό. Μια παρένθεση εδώ πρόεδρε να πω ότι μας κάνει εντύπωση γιατί απορρίφθηκε η επίσκεψη στο Μεξικό, γιατί το Μεξικό είναι ο παγκόσμιος πρωταγωνιστής, παγκόσμιος λέγω, στο εμπόριο με την κοκαίνη. Να πάμε Στι Ηνωμένε Πολιτείε λέει να μιλήσουμε με την ΤΕΑ. Την ΤΕΑ, την Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών για τα Ναρκωτικά, την μπορούμε να τη δούμε και στο Βέλιο και στη Μαδρίτη και όπου θέλετε. Διαμαρτύρομαι εντόνω γιατί απερίφθη η επίσκεψη στο Μεξικό και παρακαλώ να γραφεί στα πρακτικά. Κλείνει η παρέθεση. Τα καρτέλ στο Μεξικό λοιπόν δυσκολεύονται στο τράνζιτ. Ε, μέχρι τώρα έρχονταν από τον ε, Ατλαντικό στην Ισπανία και ε, στην Πορτογαλία. Εκεί τους κόψαν το δρόμο και πάνε στο Λίβερπουλ τώρα. Ε, τα περίφημα καρτέλ αυτά που λέγονται ΣΕΤΑΣ και είναι Επειδή λοιπόν η Ιβηρική είναι πολύ επικίνδυνη, έχουν μεταφερθεί στο Λίβερπουλ. Η Σιναλόα και η ΣΕΤΑΣ. Και η μεγαλύτερη δραστηριότητα ε, όμως τη διακίνηση παραμένει στην Ιβυρική Χερσόνησο. Αυτό οδήγησε σε ένα βίο πόλεμο που το γνωρίζετε μεταξύ των εγκληματικών αυτών ομάδων Σιναλό και Σέτας. Είναι φίλιος αδελφοκτόνος πόλεμος και αρκεί να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Καλτερών είχαν 50.000 νεκρούς στο Μεξικό. 50.000! με αποκεφαλισμούς και πάρα πολύ βίαιες ε, δολοφονίες, ε, γιατί είναι και παραστρατιωτική μέσα σε αυτά τα καρτέλ των ΣΕΤΑΣ. Ε, άλλη καινοτομία ή άλλο νέο, αυτά τα καρτέλ Σιναλόα και ΣΕΤΑΣ λοιπόν του Μεξικού, έχουν φτάσει στο Παλέρμο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια διακίνησης και διαμετακόμισης. Από χρόνο πώς θα πάω, α, πάρα πολύ άσχημα. Λυπάμαι λοιπόν που δεν προλαβαίνω να τα πω. Να σας πω τελειώνοντας τα εξή τρία. Πρώτον, στην Ιταλία το πρόβλημα είναι στην Τράγκετα και στην Καμόρα, στα χέρια αυτών, αλλά ε, λειτουργούν κυρίως μέσα ε, από το Παλέρμο, το λιμάνι. Και επίσης το δεύτερο που θέλω να πω, που έχει σχέση με όλα αυτά, η Λετωνία με το ε, ε, είναι σημερινό και οι Hells Angels και κάποιες άλλες τέτοιες συμμορίες μηχανοκίνητες μηχανοβίων διακινούν ναρκωτικά στη Δανία και όχι μόνο ναρκωτικά και ε, πνευματόδη και άλλα τέτοια ε, είδη. Πρέπει να σας πω λοιπόν το τρίτο, ότι στην Ανατολική Μεσόγειο ε, από τη διόρυγα του Σουέζ, τον Εύξηνο Πόντο και την Οδυσσό είναι μια νέα οδός που αυξάνεται και για τη διακίνηση της κοκαίνης. Η διακίνηση της Ένωσης της κοκαίνης μάλλον, ε, ε, θα αλλάξει γιατί αυξάνεται πάρα πολύ η ε, κατανάλωση πλέον στη Ρωσία και στην Ασία παρακαλώ. Έχω να πω και άλλα πάρα πολλά πρόεδρε. Ε, υπάρχουν ε, ζητήματα αλλά και κάποια άλλα που είναι θέματα αστυνομικά και εμπιστευτικά. Ευχαριστώ. Θα τα πείτε μετά όταν θα απαντήσετε, λέει ο Πρόεδρος, τα υπόλοιπα. Αν θέλετε να πείτε και άλλα που δεν προλάβατε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και ψηφίματα, ψηφίσματα για χώρες όπως είναι η Γουινέα Μπισάου και άλλες χώρες στην Αφρική που λέγουν ότι ε, μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα ε, και βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η γεωγραφική εξάπλωση και η οδή από τη Λατινική Αμερική και σε περιοχές της Αφρικής και της Ευρώπης. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιάλα Σέντερ για να μας παρουσιάσει το έγγραφό της για το τράφικινγκ. Εγώ πιστεύω ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κείμενο, παρότι είχαμε συγκεκριμένες προθεσμίες. Η πρόσφατη οδηγία και η στρατηγική δηλαδή της Κομισιόν για να μπορέσει να καταπολεμήσει την σωματεμπορία και αυτό μετά από δράση του Κοινοβουλίου μου επιτρέπουν να σας αναφέρω μερικά σημεία τα οποία σήμερα είναι απαραίτητα. Ευχαριστώ την κυρία Βασιλιάδου που είναι η συντονίστρια ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και την ε, διακίνηση ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα και η κυρία Βασιλιάδου κάποια στιγμή να συμμετέχει εδώ σε αυτήν την Επιτροπή, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτά τα οποία έχει να μας διηγηθεί είναι σαφώς πληροφο... ενημερωμένη πληροφόρηση και πολύ σημαντικά. Εγώ έχω πέντε σημεία να αναφέρω. Πρώτο, η ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να σταματήσουμε την σώματεμπορία για είτε πρόκειται για εργασιακή χρήση είτε σεξουαλική χρήση. Αυτό υποθέτει φυσικά και το μη εκμετάλλευση των ανηλίκων ή ατόμων που του στρατολογεί ή το οργανωμένο έγκλημα. Διότι πολλές φορές τα ίδια τα θύματα, από ορισμένα δικαστικά συστήματα, θεωρούνται ότι είναι ένοχοι ενώ στην πραγματικότητα είναι ε, θύματα. Μιλάω εδώ για κράχτες, πορτοφολάδες και διάφορους άλλους που τους χρησιμοποιεί το οργανωμένο έγκλημα. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή στρατηγική χρηματοδότηση, αηφορία ε, και προτείνω στην προκειμένη περίπτωση για τη διακίνηση ανθρώπων που είναι κάτι το αποτρόπαιο πραγματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ξεκινήσουμε διάφορες καμπάνιες για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη, την ε, κοινωνική απόρριψη. Ορισμένες χώρες θέλουν να αποκρύψουν τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρέπει να πετύχουμε όμως αυτό το το έγκλημα να θεωρείται αξιόπινο και κοινωνικός απορριπταίο. Στις 18 ε, Οκτωβρίου που είμαστε στις παραμονές είναι η μέρα κατά των ναρκωτικών. Θα έπρεπε εμείς ε, να πετύχουμε όμως να πετύχουμε και ένα ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας. Δεύτερο σημείο, τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία λείπουν. Η δυνατότητα να έχουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο αυτών των στοιχείων θα μας βοηθούσε στην εναρμόνιση αυτών των στοιχείων. Διότι σήμερα παρά τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μιλάμε με στοιχεία κατεκτήμηση. Δύσκολο λοιπόν εμείς να καταπολεμήσουμε ένα έγκλημα για το οποίο δεν έχουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία ή τα νούμερα είναι εντελώ διαφορετικά μεταξύ τους. Τελευταίο σημείο είναι η προστασία και η βοήθεια των θυμάτων Τώρα τα στοιχεία που έχουμε είναι στοιχεία θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε της πρώτης γενιάς, διότι αυτά τα στοιχεία μας τα δίνει μόνο το ίδιο το θύμα. Χρειάζεται Χρειάζεται λοιπόν προστασία των μαρτύρων, διότι αυτοί οι μάρτυρες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, οπότε δεν μπορεί κανείς να τους αφήνει εκτεθειμένους στους κινδύνους. Χρειάζεται προστασία αυτών των μαρτύρων. Τώρα, πρέπει να έχουμε τα μέσα και να καταφέρουμε να βρούμε άλλες φόρμουλες για να πετύχουμε την καταδίκη των εμπόρων ναρκωτικών. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εισαγγελείς, με τα δικαστήρια, διότι ναι μεν η αστυνομία διαπιστώνει ποιες είναι οι ενδυνάμοι μαφίες, πάντοτε μάλλον βλέπουμε από το 2010 και μετά να μειώνονται οι καταδίκες. Βλέπουμε ότι η αστυνομία κάνει τις έρευνές της, γίνονται οι ανακρίσεις, διαπιστώνουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο, ένα σοβαρό έγκλημα μπροστά μας και όταν έρχεται η ώρα της καταδίκης είναι πολύ μικρή. Κυρία Γιάλα Σέντερ τελειώνεται. Τελειώνω. Χρειάζεται λοιπόν με τους εισαγγελείς συνεργασία. Τελευταίο. Εξωτερική δράση. Πρόκειται για ένα δίκημα κυρίως διασυνοριακό. Χρειάζονται συμφωνίες με χώρες σαν την Κίνα, το Βιετνάμ. Πρέπει στη ρίζα να καταπολεμήσουμε το σωματεμπόριο. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σέντερ. Λαμβάνουμε υπόψη μας ε, αυτή την, ε, το αυτό το αίτημα που υποβάλλατε να το εξετάσουμε στην Επιτροπή μας κάποια στιγμή. Ακούσαμε τον κύριο Δεμέρα για τα καρτέλ των ναρκωτικών. Τώρα πάμε εμείς στην διέγκλημα... Στο θεματικό έγγραφο της Έμας Μακλάρκιν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας αυτό το θέμα του κυβερνοεγκλήματος και ευχαριστώ όσους με βοήθησαν στην έρευνά μου. Συνεχώς και περισσότερο αναγνωρίζεται το θέμα του κυβερνοεγκλήματος και είναι ουσιώδες να το εξετάζουμε και εμείς συχνά για να ενημερωνόμαστε. Τώρα σε λίγο θα γίνει ένα σεμινάριο για τη συνεργασία των χωρών μελών κατά του κυβερνοεγκλήματος και αυτό το μήνα στη Βουδαπέστη έγινε μια διάσκεψη που ήταν η δεύτερη του είδους της μετά την σχετική του Λονδίνου. Σχεδόν 600 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, επιστημόνων και απλών ανθρώπων, δηλαδή κοινωνίας των πολιτών πήγαν εκεί. Καθώς και οργανώθηκε και ένα βήμα για τους νέους ειδικά. Αυτόν το μήνα επίσης πάνω από 300.000 επιχειρήσεις στο διαδίκτυο ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καταπολεμηθεί το κυβερνοέγκλημα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για το συντονισμό όλων αυτών των προσπαθειών. Παραπάνω από κάθε άλλο είδος οργανωμένου εγκλήματος αυξάνεται πολύ γρήγορα το κυβερνοέγκλημα. Ελπίζω το έγγραφό μου να σας δείξει πόσο πολλές και διαφοροποιημένες είναι οι λειτουργίες του κυβερνού εγκλήματος και πόσο ουσιώδης θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ένωσης για την καταπολέμησή του. Μπορεί να μας αφορά όλους, να μας κλέβει την ταυτότητά μας και να παράγει ή να πουλάει μάλλον ε, φάρμακα μαϊμούδες και να δημιουργεί και κυβερνοϊούς που βλάπτουν όλων μας τους υπολογιστάς. Μπορεί επίσης να αποτελέσει φυτόριο τρομοκρατών και να οργανώσει επιθέσεις κατά πληροφορικών συστημάτων ολόκληρων. Τέλος, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό ή τόσο καλά οργανωμένο από χρηματοδοτικής απόψεω. απόψεως. Επομένως το καθήκον μας είναι να τονίσουμε τη σημασία που έχει η συνεργασία για την αντιμετώπιση του και η γνώση των πολιτών περί του κινδύνου. Η επιμόρφωση πρέπει να αρχίσει από τους τόπους εργασίας και να φτάσει μέχρι τα σπίτια. Πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι κάθε φορά που κατεβάζουν ένα βίντεο ή ένα τραγούδι που δεν έχουν πληρώσει μπορεί τελικά να χρηματοδοτούν και το οργανωμένο έγκλημα έτσι. Όποτε αγοράζουν ένα φάρμακο από το ίντερνετ μπορεί να θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Και όποτε που έχουν πρόσβαση σε άλλον υπολογιστή χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εγγυήσεις μπορεί κάποιος να τους εκμεταλλευτεί. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και εμείς και η Ευρώπη γενικότερα. 388 δισεκατομμύρια δολάρια κοστίζει το κυβερνοέγκλημα σε όλους μας κάθε χρόνο. Το ενθαρρυντικό είναι ότι το μήνυμα αυτό αρχίζει να ακούγεται και συγχαίρω την Ευρωπόλ που έχει μία ομονάδα ειδική καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος καθώς και την Κομισιόν για την σύνταξη της τελευταίας της οδηγίας για το θέμα. Καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να το λύσει. Η συνεργασία με κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα πρέπει να θεωρείται κάτι το στοιχειώδες και προτεραιότητα για τη διεθνή διπαλωματία, διότι το ίντερνετ βέβαια δεν σταματάει στα σύνορα της Ένωσης, είναι παγκόσμιο και τα προϊόντα λογισμικού πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους τον κίνδυνο που μπορεί να εμπεριέχει η χρήση τους και να προσπαθήσουν όλοι μαζί να προβλέψουν τις συνέπειες. Η Ευρωπόλη, η Ιντερπόλ, το ΝΑΤΟ και το FBI όλοι συνεργάζονται για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και πρέπει να εναρμονιστούν οι ποινές και οι κυρώσεις που προβλέπονται πανενωσιακώς. Πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους σε όλα αυτά και να δημιουργήσουμε προβλήματα, ε, προγράμματα επιμόρφωσης και για τους πολίτες. Δεν είναι εύκολο βέβαια, αλλά νομίζω ότι εδώ πρόκειται για θέμα όπου αν τα καταφέρουμε θα έχουμε κάνει κάτι σημαντικό και τονίζω ιδιαίτερα τη σημασία να παραμείνει η προτεραιότητά μας το θέμα για να διασφαλιστεί δε η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών και καταναλωτριών δεν πρέπει να φοβόμαστε να επιδείξουμε ιδιαίτερο θάρρος. Αλλιώς δεν θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα όπως πρέπει. Σας κατευχαριστώ. Ο συνάδελφός μας Γκέι Μίτσελ έχει έρθει να παρουσιάσει το δικό του έγγραφο. Σε σχέση με τη δίμευση των περιουσιακών στοιχείων και τις κατασχέσεις γενικότερα ως τρόπο αντιμετώπισης, ε, θα κάνετε και εσείς την παρουσίασή σας και μετά ε, οι συνάδελφοι για να μπορέσετε να απαντήσετε στη συνέχεια. Και αν δεν μπορέσετε στην πρώτη σας τοποθέτηση να ολοκληρώσετε, έχετε και δευτερολογία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πάω να ψηφίσω. Στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Ελπίζω λοιπόν να προλάβω και το τέλος της συζήτησης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το έγγραφο. Ο βασικός στόχος είναι να τονίσουμε την ανάγκη ενός ε, μοντέλου κατάσχεσης προϊόντων εγκλήματος σε όλη την ε, Ευρώπη. Ο ΙΕ έχει υπολογίσει σε 2,1 εκατομμύρια δολάρια ή 3,6% του παγκοσμίου ΑΕΠ το προϊόν εγκλήματος παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν ε, τέτοια στοιχεία σίγουρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα είναι δισεκατομμύρια τα κέρδη γιατί ενδιαφέρομαι εδώ εγώ γι' αυτό, γιατί η χώρα μου Ιρλανδία έχει ένα πολύ προηγμένο σύστημα, μοντέλο που βασίζεται στο αστικό δίκαιο και είναι σημαντικό να μοιραστούμε την εμπειρία μας. Τον Ιούνιο του 1996 ένας αστυνομικός μας κυβερώνει η μια δημοσιογράφος ερευνητικής ε, δημοσιογραφίας δολοφονήθηκαν από μια εγκληματική οργάνωση, οργανωμένο εγκλήματος. Και αυτό ήταν καταλήτης για την πολιτική βούληση να υπάρξει ένα ε, σωστό μοντέλο και σύστημα κατάσχεσης προϊόντων εγκλήματος. Μέσω φόβου ή οικονομικής πίεσης ε, διέφευγαν και έμειναν ατιμόρυτοι αυτοί οι εγκληματίες μέχρι τότε. Τώρα με αστικές διαδικασίες στο δικαστήριο, χωρίς πρώτερη καταδίκη σε ποινικό δικαστήριο, μπορούμε να κατάσχουμε το προϊόν εγκλήματος. Για να δημιουργηθεί λοιπόν ένα πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να βοηθήσουμε και να δημιουργηθούν ε, σημαντικές δομές. Χρειάζεται βεβαίως περισσότερη δουλειά για να έχουμε ένα συγκεκριμένο κοινό σχήμα και σύστημα κατάσχεσης. Ε, εγώ αναφέρω τα διάφορα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στην ε, Ιρλανδία, συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ε, μεταξύ των αντιστοίχων υπηρεσιών κατάσχευσης και ένα δίκτυο και διάφορα μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποια στοιχεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, είναι μια πρώτη νομοθετική πρόταση και η επόμενη Ιρλανδική Προεδρία θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι θα τεθούν διάφορα ζητήματα όμως μέχρι να τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία και να μπορέσει να εφαρμοστεί. Παράδειγμα, το πεδίο εφαρμογής ε, τι θα γίνει ας πούμε με το πάγωμα και τη δίμευση και τα αντίστοιχα ε, ε, εντάλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει προηγηθεί ποινική δίκη για να μην πω καταδίκη. Αυτό είναι δύσκολο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τα νομικά συστήματα και την ένωμη τάξη της κάθε χώρας. Υπάρχουν θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα που αναπόφευκτα θα τεθούν από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος. Θα μπορούσε και πάλι όμως η Ιρλανδία να αποτελέσει μια προηγούμενη ε, κατάσταση και να δείξει πώς μπόρεσε να λύσει αυτά τα θέματα στη χώρα. Υπάρχει το άρθρο 6 βεβαίως Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τη δίκαιη δίκη, για την προστασία και αντίστοιχα πρωτόκολλα. Και το άρθρο 7 ε, ας πούμε της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τέλος, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι βασικός στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προσφέρει στους πολίτες ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα με ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και προσώπων δεδομένη σε συνδυασμό με την πρόληψη εγκλήματος. Στη συνθήκη της Βόνας αυτό είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα θέματα εσωτερικών και δικαιοσύνης. Θα πρέπει αυτό να το αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε προς όφελος των πολιτών και να μην μπορούν να ξεγλιστρούν και να ξεφεύγουν οι εγκληματίες, να φεύγουν από τη μια χώρα στην άλλη και να γλιτώνουν, να μένουν ε, ατιμόρυτοι. Να έχουμε ένα κοινό σύστημα με κοινέ τιμωρίε και αυτό θα είναι προ όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μίτσελ και όλους τους ε, συντάκτες και των τεσσάρων θεματικών εγγράφων καθώς επίσης και τον κύριο Γιακολίνο για το δικό του έγγραφο. Έχουμε μια ανάλυση έτσι, αρκετά συνολική της κατάστασης, αλλά και λεπτομερής. Και σε παραδοσιακούς τομείς οργανωμένου εγκλήματος, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η διακίνηση ανθρώπων, αλλά και νέους τομείς όπως το κυβερνοέγκλημα και βεβαίως δυνατότητες δράσης, η δίμευση και κατάσχεση περιουσιαστικών ε, στοιχείων ε, και προϊόντων εγκλήματος που πρόκειται για δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπατε, κάθε χρόνο. Και έχουμε και οικονομική κρίση. Δεν έχουμε προβλέψει να μιλήσουν οι συντονιστές ε, ξεχωριστά και μετά τα μέλη. Δεν ξέρω τι θέλετε. Έχουν ζητήσει το λόγο κάποιοι συνάδελφοι η κυρία Γιαννάκου και η κυρία Καβριέλ. Δεν ξέρω άλλοι. Αν δεν διαφωνούν οι συντονιστές, αμέσως τα μέλη. Παρακαλώ κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, πραγματικά είναι αξιόλογες οι συμβολές και του εισηγητού φυσικά και των τεσσάρων συναδέλφων. Ιδιαίτερα ε, σημαντικό είναι αυτό που σημειώνει ο εισηγητής κάνοντας προτάσεις φέρνοντας στο προσκήνιο τον Ιταλικό νόμο για την διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων ε, και κυρίως αυτό που έχει σημασία, το να μην μπορεί οποιοδήποτε να διαφεύγει σε άλλη χώρα όπου το νομοθετικό πλαίσιο είναι είτε ευέλικτο είτε πολύ ελαστικό. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Παρακολουθώντας την ε, διαδρομή, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και υπήρξα παλιά πρόεδρος της Επιτροπής έρευνας για τα ναρκωτικά, παρακολουθώντας την πορεία των πραγμάτων από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα, πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα. Εάν εξαιρέσετε τη συμβολή ε, προσώπων από τις ανατολικές χώρες ε, μετά το άνοιγμα και μετά την κατάρρευση του τείχους και τις ομάδες, ε, τις εγκληματικές οργανώσεις που έχουν δημιουργηθεί εκεί ε, πρέπει να σας πω ότι και τότε τα λιμάνια όχι μόνο της Ιβηρικής, το Άμστερνταμ και το Λίβερπουλ ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικά, η Νιγηρία και οι χώρες της Δυτικής Αφρικής και βέβαια είναι επιβεβαιωμένη η σχέση της τρομοκρατίας με το εμπόριο των ναρκωτικών μιλώντας για, το, ε, για την έκθεση του συναδέλφου για τα ναρκωτικά. Επομένως δεν τίθεται ερώτημα όπως αναφέρει στο τέλος της έκθεσης του. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Και αναφέρεται και σε δική μου έκθεση του 1987 για το εμπόριο κοκαίνης στη Λατινική Αμερική. Όπως είναι επιβεβαιωμένη η καλλιέργεια ηρωίνης στη Λατινική Αμερική από μεγάλες επιχειρήσεις που έκαναν ξέπλυμα χρημάτων. Επειδή αναφέρθηκε ο συνάδελφος στην DAE, θέλω να σημειώσω ότι δεν έχει καμία σχέση η πληροφόρηση που θα μπορούσε να πάρει κανείς στη DA στη Ουάσιγκτον μέσω του Γενικού Διευθυντού και των στελεχών με αυτά που μπορεί να μάθει στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Καμία σχέση. Οι βασικές πληροφορίες για το πώς κινείται το πράγμα σήμερα... Κύριε Πρόεδρε, με διακόπτη, δεν καταλαβαίνω. Εγώ κάνω τις παρατηρήσεις μου. Συγγνώμη, ε, το αντίθετο είπα ότι... δεν χρειάζεται να πάμε στι Ηνωμένε Πολιτείε για να δούμε την Δία. Θα τη δούμε και στην Ευρώπη. Αυτό είπα. Συγγνώμη να το διευκρινίσω. θα ήθελα να το διευκρινίσω. Ήθελα να πω ε, ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δύο λεπτά ο καθένας ε, έχετε. Παρακαλώ ολοκληρώνετε. Και θέλω να πω και στον κύριο Μέρα κάτι. Κύριε Ντίας Δεμέρα, μη διακόπτη παρακαλώ. ένα ταξίδι στις ε, από λίγου ανθρώπους από την Επιτροπή μας για να δουν το Γενικό Διευθυντή του, της DA, το Γενικό Διευθυντή του FBI και βέβαια στην Ευρώπη πρέπει να δούμε το Γενικό Γραμματέα της Interpol ε, ε, ο οποίος έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες από όλους τους υπόλοιπους για να κρίνουμε ποια νέα μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι είναι προϊόν ανθρώπινη δραστηριότητα το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, όλα αυτά και το πάση φύσεω έγκλημα. Αλλά και προϊόν ανθρώπινη δραστηριότητα είναι η καταπολέμησή του. Είναι φανερό ότι τα τελευταία χρόνια τρέχουμε πίσω από το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να βρούμε πιο έξυπνου, πιο ευέλικτου τρόπου σε όλα τα επίπεδα και στη δικαιοσύνη και στην καταστολή για να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον ένα μέρος από αυτές τις δραστηριότητες γιατί όλες δεν νομίζω ότι φαντάζεται κανείς ότι μπορεί να συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αντιπροσωπείες εκτός ενώσεως ε, θα συζητηθούν στη συνεδρίαση των συντονιστών και όχι εδώ. Ε, μετά, η κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και τους τέσσερις συναδέλφους. Ήταν πάρα πολύ εύστοχα αυτά που είπαν. Αν δούμε και τα τέσσερα ε, έγγραφα μαζί, μπορούμε από τώρα να σκεφτούμε κάποιες κοινέ συστάσεις που είναι και απαραίτητες, αλλά και πρέπει να απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής για τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Θέλω να αφαιρθώ περισσότερο στο έγγραφο της κυρίας Αγιάλα για τη διακίνηση ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό εδώ στην Επιτροπή μας να δώσουμε και να έχουμε και την άποψη της κυρίας Βασιλιάδου, να την ακούσουμε, γιατί κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ενέργεια, είναι πολύ δραστήρια και έχει πάρα πολλές προφορίες και δεν μπορώ παρά να υποστηρίξω την πρόταση της κυρίας Αγιάλα. Να έρθει η κυρία Βασιλιάδου να μας τα πει. Επίσης, θέλω να κάνω μερικά σχόλια. Είναι οπωσδήποτε σημαντικό να συνεχίσουμε να επιμένουμε για την πρόληψη εκστρατείες, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης να οργανώνουμε για ένα φαινόμενο που είναι τόσο σοβαρό και τόσο περίπλοκο και βαρύ. Μετά, για την εκπαίδευση των αστυνομικών και των άλλων υπαλλήλων, των άλλων υπηρεσιών θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκπαιδευμένοι για να μπορούν να αναγνωρίζουν ε, το τράφικινγκ καμιά φορά γιατί είναι και ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολλά πλοκάμια και διαφοροποιείται με τον καιρό, παίρνει νέες μορφές. Όπως γνωρίζουμε οι εγκληματικές οργανώσεις προσαρμόζονται στις εποχές. Ε, στη συνέχεια, τρίτον, πολύ συγκεκριμένη πρόταση, να έχουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό για να βοηθούμε τα θύματα. Το είπε η κυρία Γιάλα και σωστά. Σε 18 κράτη-μέλη πάνω κάτω υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, σε άλλα κράτη δεν υπάρχει. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πρόταση. Και έχω και μια ερώτηση επίσης συγκεκριμένη. Πρώτον, γιατί δεν μπορούμε ε, να αρχίσουμε από το να ταυτοποιούμε καλές πρακτικές και να τις διαδίδουμε. Μέγα έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, ποια είναι τα οικονομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και οι πόροι για να ενισχυθεί ο συντονισμός και να υπάρχουν περίφημες βάσεις δεδομένων που μας λείπουν. Παράδειγμα, τι γίνεται με τις μικτές ομάδες ε, διοκτικών αρχών που θα μπορούν να καταπολεμούν αυτό το θέμα γιατί από τη μικρή πύρα που έχουμε αποδεικνύεται ότι ε, πολύ γρήγορα γνωρίζουν τέτοια εμπόδια οι μικτές αυτές ομάδες. Θα πρέπει να ξέρουν ξένες γλώσσες για να μπορούν να συνεννοούνται. Θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν ισχύει αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή και εκεί χρειάζεται εκπαίδευση. Και ένα τελευταίο για τις εταιρικές σχέσεις και συνεργασία με διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να ενέχεται περισσότερο. από το Κοινοβούλιο να ζητήσουμε αυτές οι εταιρικέ σχέσεις και οι συνεργασίες να γίνονται πιο γρήγορα. Γιατί στη στρατηγική που μας έφερε τον Ιούνιο η κυρία Βασιλιάδου προβλέπεται κάτι τέτοιο, αλλά μόνο από το 2014. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι το 2014. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση. Και πάλι συγχαρητήρια στην κυρία Γιάλα. Έχουμε πραγματικά πολλά στοιχεία που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην αναζήτηση κοινών συγκεκριμένων προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ. Για τις προτάσεις σας η γραμματεία μου μας μου θυμίζει ότι το 2013 προβλέπονται τέτοιες συναντήσεις. Τώρα η κυρία Κοστέλου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τους τέσσερις εισηγητές και εισηγητρίες για τα θεματικά τους έγγραφα, καθώς και τον γενικό εισηγητή. Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν μια πολύ καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση. Να κάνω μερικά σχόλια τώρα. Για τα καρτέλ των ναρκωτικών και το έγγραφο που αφορούσε το δουλεμπόριο. Νομίζω ότι ενδιαφέρον θα ήταν η δημιουργία μιας ειδική τηλεφωνικής γραμμής για τη βοήθεια των θυμάτων κατάχρησης ναρκωτικών ή δουλεμπορίου είναι πολύ θετική και γι' αυτό το τελευταίο θα ήθελα να πω συγκεκριμένα ότι μου άρεσε ιδιαίτερα το έγγραφο η συντάκτρια αναφέρει πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία και την ανάγκη να συλλέγονται τέτοιου είδους στοιχεία, δεν υπάρχουν αρκετά. Όσο για την κατάσχεση περιουσιών από εγκληματικές δραστηριότητες, το πρότυπο που ισχύει στην Ιρλανδία είναι πολύ καλό. To support the suggestion um, διότι σε αυτό το, κατά αυτό, σύμφωνα με αυτό το πρότυπο γίνεται επανεπένδυση των κατασχεθέντων στοιχείων για κοινωνικούς σκοπούς. Υπάρχουν βέβαια κοινά θέματα για όλα τα έγγραφα, όπως για το κυβερνοέγγριμα, έτσι και για τα άλλα υπάρχει το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης Έχω και μερικά ερωτήματα. Γενικά για τα έγγραφα είναι εξαιρετικά, τα συμπεράσματα ενδιαφέροντα, αλλά Εσύ να μας, εσείς να μας πείτε κύριε Πρόεδρε, πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά για να έχουμε τελικά μία κάποιο αποτέλεσμα. Καλά είναι τα έγγραφα, αλλά θέλουμε να δούμε και πώς θα δράσουμε, πώς θα μεταφράσουμε όλα αυτά σε δράση. Thank you, Mrs. Costello, and, uh, Ευχαριστούμε κύριε Κοστέλου. Επειδή είχατε συγκεκριμένα ερωτήματα, ας απαντήσουν οι συντάκτες. Έχουμε όμως πρώτα ακόμα έναν για αυτόν το γύρο και επειδή εσείς ψηφίζετε στην εικόνα και μπορεί να χρειαστεί να φύγετε νωρίτερα, όταν τελειώσει ο γύρος να ξαναμιλήσετε. Τώρα για το περιεχόμενο των θεματικών εγγράφων και για το γενικότερο του κυρίου Γιακουλίνο, όλα αυτά, όλα αυτά λέγω, θα δουν πρώτα οι συντάκτες και τις τροπολογίες και θα συνδυαστούν από τον Γενικό Εισηγητή. Στην τελική έκθεση στα τέλη του 13 μάλλον, αν εγκριθούν από τους συντονιστές και συντονίστριες βέβαια τα χρονοδιαγράμματα. Η κυρία Βάιλερ λοιπόν τελευταία σε αυτόν τον γύρο και μετά ο κύριος Γκέι Μίτσελ. Κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εγώ μια πολύ συγκεκριμένη και μικρή τοποθέτηση έχω. διότι δεν μπόρεσα να μελετήσω σε όλες τις λεπτομέρειες το έγγραφο για κολίνο. Από αυτά που διάβασα όμως πρέπει να σας πω ότι τα βρίσκω πολύ διαφωτιστικά και πολύ χρήσιμα για τη δουλειά μας και πραγματικά τώρα κάναμε μια τομή. Όλα αυτά που έχουμε μάθει μέχρι σήμερα τα έχουμε επεξεργαστεί και τα συζητούμε εδώ. Λοιπόν, ας τα κοιτάξουμε, ας τα αξιολογήσουμε σε μια πρώτη φάση Σήμερα το πρωί που εγκαινιάσαμε ε, έτσι πανηγυρικά ε, τη βδομάδα για τα 20 έτη της ενιαίας αγοράς διαπιστώνουμε πόσα έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έρχομαι τώρα εδώ και βλέπω πόσα λίγα έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα έχει καλές ιδέες και πρακτικές Ας πούμε στο ε, ίδιο κράτος σε μία επικράτεια είναι ενιαίος ο αριθμός κλήσης, αλλά μπορεί το διπλανό κράτος να μην γνωρίζει καν ότι υπάρχει τηλεφωνικός τέτοιος αριθμός. Και πουθενά αυτά δεν συλλέγονται, ούτε ε, καταγράφονται, ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν απατώμε. Υπάρχει τέτοια μονάδα που να ασχολείται με αυτό το θέμα που είναι για μας ε, χρήσιμο. Ας πούμε, στην Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς, στην ΙΜΚΟ, εγώ ασχολούμαι και προβληματίζομαι με τα θέματα απάτης, ε, ιδιαίτερα στις δημόσιες συμβάσεις. Και λέτε εδώ και πολύ σωστά το λέτε κυρία Κολίνο στα συμπεράσματα ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και διανόμου και την πρόταση Ταραμπέλα, να λέμε ότι εταιρείε που καθιοδήποτε τρόπο έχουν τραβήξει την προσοχή λόγω εγκληματικών δραστηριών να αποκλείονται από τις ε, συμβάσεις και τους διαγωνισμούς. Αυτό δεν είναι καινούριο, αυτό υπάρχει ήδη. Αλλά θα πρέπει να δούμε. Βέβαια δεν μιλάμε για τα μικρά ψάρια τώρα, αλλά τα μεγάλα ψάρια φορά ε, και εκατομμύρια διακινούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στις δημόσιες συμβάσεις. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε πάντα στο δικαστήριο ε, και ποια περίπτωση συζητούν γιατί δεν φτάνουν πάντα αυτές οι υποθέσεις στο δικαστήριο. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε μια μονάδα συντονισμού, κάπου μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που να συλλέγει αυτά τα στοιχεία και να ανταλλάσσουμε και εμπειρίες. Τι έχει γίνει, τι ισχύει και στην επόμενη μελέτη αντικτύπου να τα βάζουμε και αυτά στην αξιολόγηση. Ε, όπως σας είπα, έχουν γίνει πολλά σε, εθνικό επίπεδο, λίγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν γνωρίζει η αριστερά τι πει η δεξιά, όπως λέμε στα γερμανικά. Και αυτό είναι ε, καθήκον του Κοινοβουλίου του ίδιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάιλερ. Ωραία. Τώρα ακολουθούν οι απαντήσεις των συντακτών των εγγράφων. Είναι πάρα πολύ λεπτομερή τα έγγραφα και πολλές πληροφορίε, πληροφορίες, στατιστικές και τα στοιχεία. Ορισμένα τα ακούμε για πρώτη φορά εδώ στην Ειδική Επιτροπή, ιδιαίτερα τα όσα λέγει το έγγραφο της κυρίας Αγιά Λασέντερ, ο αριθμός των ατόμων, που υποχρεώνονται σε καταναγκαστική εργασία. υπολογίζονται περίπου σε 900.000, περίπου ένα εκατομμύριο και 270.000 υφίστανται σεξουαλική εκμετάλλευση. Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μίτσελ που πρέπει να πάει να ψηφίσει σε άλλη επιτροπή για να απαντήσει σε ερωτήσεις που του έγιναν για το έγγραφό του, για την κατάσχεση των προϊόντων εγκλήματος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με διευκολύνετε να πάω να ψηφίσω. Για πρώτος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τον κύριο Γιακολίνο και τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους για τη γενική συνεργασία. Το εκτιμώ πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ να μπορώ να συνεργάζομαι με συναδέλφους με αυτόν τον τρόπο. Και για τις ερωτήσεις σας ευχαριστώ. Συμφωνώ να χρησιμοποιούνται για κοινοφελείς σκοπούς ε, αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαμε να δούμε τα προηγούμενα. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να καθορίσουμε κατευθυντήριες γραμμές. Σας είπα αν ενδιαφέρεστε στην Ιρλανδική Προεδρία. Ε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι εξέχον δικηγόρος και ενδιαφέρεται ε, να προωθήσει αυτό το θέμα. Αν θέλετε και αν σας ενδιαφέρει να τον καλέσουμε στην Επιτροπή μας να είναι χρήσιμο και για τον ε, εισηγητή μας και για την πρόεδρο, θα πρέπει να αντεπιτεθούμε, όχι μόνο για να το νιώσουν στο πετσί τους οι εγκληματίες, αλλά να δει και η κοινή γνώμη ότι κάποιος τιμωρείται, ότι δεν ξεφεύγουν έτσι ατιμωρητοί, ότι αποδίδεται δικαιοσύνη πραγματικά. Και όταν κάποιος έχει τεράστια περιουσία, χωρίς να έχει δουλέψει ποτέ ή δεν έχει δουλέψει τελευταία δεκαετία ας πούμε, θα πρέπει να του ζητούνται οι λόγοι και το πόθεν έσχεσαι. Αν μπορεί να τα δικαιολογήσει, ωραία. Δεν θα δώσει συνέχεια ούτε θα διωχθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν όμως δεν μπορεί, στην Ιρλανδία θα πάμε και θα πούμε, εσύ έχεις 10 εκατομμύρια στην τράπεζα, έχεις αγωνιστικό ε, αυτοκίνητο, φόρμουλα 1, ξέρω εγώ, και πού τα βρήκες όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω, αυτά μπορούν με εντάλματα αστικού δικαίου να κατασκεθούν, χωρίς να έχει προηγηθεί η ποινική δίκη και η καταδίκη. Στη συνέχεια, εγώ γνωρίζω το Ιρλανδικό παράδειγμα, αλλά αυτά τα κάνουν οι διοκτικές αρχές, η αστυνομία μας, ε, ε, η εφορία, η ακτοφυλακή, το λιμενικό και άλλες υπηρεσίες. Στην αρχή ανησυχούσαμε πολύ. Τι θα κάνει η αστυνομία, μπορεί να πάει ε, στην κοινωνική ασφάλιση, στην εφορία, να πάρει στοιχεία, τι τους νοιάζει, δεν επικοινωνούν. Ε, υψωνόταν ένα συνικό τείχο. Σου λένε «Ε, εδώ προστατεύεται ο κόσμος, υπάρχουν θεμελιώδη δικαιώματα. Και όμως αυτή η προσπάθεια ευωδόθηκε, δικαιώθηκε και ε, πραγματικά συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και μπορούμε να προχωρήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται βεβαίως κάπως να περιστούν οι πολιτικές ευθερίες, δεν αντιλέγω, αλλά θα πρέπει να δούμε πού έχουν λειτουργήσει καλά. Δεν είναι μόνο η Ιρλανδία, είναι και άλλες χώρες που το κάνουν. Και θα πρέπει να το προωθήσουμε και το Συμβούλιο Υπουργών μπορεί να πιστεί, γιατί η Κομισιόν έχει ήδη πιστεί. Είναι σημαντικό εμείς ως θεσμικό όργανο κλεγμένο από τους λαούς να το υποστηρίξουμε επί της αρχής. Τις λεπτομέρειες βεβαίως θα τις δούμε αργότερα, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο βήμα προς τα εμπρός. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα με την κανονική σειρά, ο ε, συνάδελφος Δίας Δεμέρα, θα προτείνω να χρησιμοποιήσουμε ως Ε, χρονικό πλαίσιο ε, την τοποθέτηση του κυρίου Γκέι Μίτσελ που μίλησε τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ να μην υπερβείτε το τετράλεπτο και εσείς οι υπόλοιποι. Ο κύριος Δίας Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο δηλώσεις. Εγώ τρέφω απόλυτη εμπιστοσύνη στις διερμηνευτικές ικανότητες των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τα τζάμια. Ε, και διαμαρτύρομαι γι' αυτό, γιατί για να μιλήσει κανείς με την Δία δεν χρειάζεται να πάει στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εμείς θα λάβουμε περισσότερες πληροφορίες από τις ε, Δία ε, στην Ευρώπη από ότι τις Αμερικάνικες. Εγώ φαντάζομαι από τη Λιόνι από τη Μαδρίτη θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες η δεύτερη δήλωση σχετικά με το θέμα του Λίβερπουλ Αυτό το λέω στο κείμενό μου, φτάνει να το διαβάσει κανείς. Το θέμα του Λίβερπουλ δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Δεν ήταν απλώς η αναζήτηση εναλλακτικών οδών ε, πρόκειται για ένα ε, εκ νέου φαινόμενο, δηλαδή υπερπόντιες βάσεις. Όχι μόνο λαμβάνουν, αλλά πάνε και την ψάχνουν. Ε, ευχαριστώ. Εγώ να σας πω ότι εμείς έχουμε μια μόνιμη αντιπροσωπεία στη Ουάσιγκτον, στην οποία μπορεί κανείς να απευθυνθεί για να λάβει πιθανές πληροφορίες που μας χρειάζονται. Είναι η μόνη μας, η μόνη μας μόνιμη αντιπροσωπεία στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πάω τώρα στην κυρία Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη, αλλά κυρίως για τις διευκρινήσεις που έγιναν ε, για το έγγραφο. Ευχαριστώ και το, τη γραμματεία της Κομισιόν και για την ε, τεράστια υπομονή που είχε ο άνθρωπος για να με βοηθήσει. Συμφωνώ απόλυτα ότι χρειάζεται πρόληψη. Εμείς θα πρέπει να έχουμε πρόληψη, όχι μόνο όταν έχουμε πια τον δρόμο που έχει ακολουθήσει το χρήμα να προχωράμε στην κατάσχεση κλπ. κλπ αλλά να μπορούμε να διαπιστώσουμε εν γενέση από τον τραπεζικό λογαριασμό. Ή υπήρχαν ας πούμε γραφεία τα οποία ε, ναυτιλιακά γραφεία τα οποία διαχειριζόντουσαν όλη την πειρατεία στη Σομαλία. Πρέπει να πάμε να τους ψάξουμε για την κυρία Γαβριέλ. Ε, σίγουρα χρειάζεται κατάρτιση και καλές πρακτικές. Βέβαια ελπίζουμε την οδηγία να την εφαρμόσουν όλα τα κράτη ταυτόχρονα. Αυτό θα βοηθήσει να μειώσουμε την σωματεμπορία για σεξουαλικούς και εργασιακούς λόγους. Τα νούμερα είναι πραγματικά σκανδαλώδη. Και πρέπει να ενισχύσουμε και το ανθρώπινο δυναμικό. Το θέμα των εκστρατιών όπως ε, γίνεται καμπάνια και λέει το τσιγάρο βλάπτει, ε, τότε θα πρέπει να γίνει και μία καμπάνια, ούτως ώστε όλοι να ενημερωθούν για το τι εστί σωματεμπόριο. Και να, υπάρχει, να ενημερωθούν επίσης αυτοί, αυτοί που θα μπορούσαν να είναι θύματα του σωματεμπορίου για αυτήν την πράσινη γραμμή, την helpline, για να μπορέσουν να προσφύγουν. Λοιπόν, και για το θέμα των ε, πόρων. Ε, δεν το έβαλα στο κείμενο, διότι το κείμενο ήδη το έκανα μακρύ σε σχέση με αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί. Λοιπόν, η περίοδος για τη λειτουργία της οδηγίας είναι 2012-2016. Εμείς δουλεύουμε ήδη για το 2020. Θα μπορούσε να έρθει η κυρία Βασιλιάδου και να μας δώσει παραπάνω στοιχεία. Να μας πει πόσο χρήμα θα πάει στην καταπολέμηση της ε, σωματεμπορίας και κλπ λέει ο Μιλήτρια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε αυτές τις ε, ε, πληροφορίες για να υποστηρίξουμε δηλαδή και το αίτημα για κονδύλια. Ευχαριστούμε. Τώρα για το κυβερνοέγκλημα η κυρία Μακλάρκιν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους όσους έκαναν σχόλια. Το κύριο όμως συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε το ίδιο γρήγορα με τη δράση των εγκληματιών οι οποίοι αλλάζουν τα πρότυπα λειτουργίας των εγκληματικών τους επιχειρήσεων γρηγορότατα, ταχύτατα. Υπάρχει βέβαια κάποια παρακολούθηση, πρέπει να τα μελετήσουμε αυτά, να δούμε τι ακριβώς κάνουν και την προσπάθειά μας να την κάνουμε χωρίς επικαλύψεις αλλά ταχύτατα. Να μάθουμε πώς, πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία υπέρ ημών. Οι εγκληματίες αυτό κάνουν. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από αυτού του θέματος και να καταλήξουμε σε πραγματικές συστάσεις με πραγματική επίπτωση. Ευχαριστούμε. Για τα συμπεράσματα ο συνάδελφός μας Γιακουλίνου. Στο, στη γενική του εισηγήση. Ορίστε Σαλβατόρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω πολλά. Στο σωστό δρόμο είμαστε. Όλες οι συνεισφορές των συναδέλφων είναι σαφείς επαναλαμβάνουμε με δύναμη ότι ο αγώνας αποτελεί προτεραιότητα των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αγώνας για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος. Εμείς σε συνεργασία με την γραμματεία πληθυντικός μεγαλοπρέπειος του εισηγητή, θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε στον κορμό του κειμένου μου όσο καλύτερα μπορούμε το κείμενο, τα κείμενα μάλλον των συνεισφορών του συναδέλφου. Και η έκθεση στα μέσα της θητείας θα εμπλουτιστεί και από τις τροπολογίες των συναδέλφων. θα ενισχύσουμε την νομοθεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. και κυρίως πρέπει να παλέψουμε για την αναγνώριση του εγκλήματος σύστασης συμμορίας για εγκληματικούς λόγους. θα έχουμε κερδίσει μία μάχη, αλλά θα έχουμε κερδίσει και ένα βήμα πολιτισμού. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, βοηθούς, γραμματεία για όλη τη βοήθεια που μας δώσανε. Κυρία Μπορσελίνο, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα διάφορο. Επειδή είναι η τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας πριν επισκεφθούμε την Ιταλία, εγώ έχω εδώ το πρόγραμμα με τις συναντήσεις. Θέλω να υπογραμμίσω ότι στις συναντήσεις μας στο Μιλάνο δεν έχουμε ραντεβού που θεωρούσαμε πολύ σημαντικά. Δεν, δεν βλέπουμε κανέναν που να ασχολείται με την ανακύκλωση του χρήματος, δεν βλέπουμε εισαγγελίες που ασχολούνται με τη διαφθορά, δεν ε, βλέπουμε και τους εκπροσώπους του Μιλάνο 2015 που είχαν μιλήσει για δίσδυση της μάπια στη δημοπράτηση των έργων για την έκθεση. Εγώ θα έλεγα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα στους συντονιστές που θα ακολουθήσουν. Πολύ σύντομα. Ε, ε. Μου λένε ότι πολλοί συνάδελφοι, μάλλον οι ερμόδιοι για τη συνάντηση αυτή δεν ήταν παρόντες, μπορούμε όμως να το συζητήσουμε στους συντονιστές. Λοιπόν, για, άλλα διάφορα, όχι. Πέρα στη συνεδρίαση, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες 12 Νοεμβρίου του 2012 από τις 3 στις 6.30. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλα διάφορα και στις 5.30 έχουμε συνάντηση συντονιστών. Δεν είναι όλοι οι συντονιστές όμως παρόντες, οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι να έρθουν όλοι οι συντονιστές. Ευχαριστώ.